Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Και ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας εκεί που σταματήσαμε το πρωί. κοιτάξουμε τις πρακτικές και δημοσιονομικές συνέπειες των διατάξεων και ρυθμίσεων που αφορούν την έδρα της ΕΝΙΣΑ, της Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Δικτύων και της Πληροφορίας. Euh, entre euh, και την, ε, θα συστήσουμε λοιπόν την Ελλάδα και την ε, κατανομή της έδρας μεταξύ Ηρακλείου και Αθήνας. Καλωσορίζω τον κύριο Έλμπρεχτ, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση δεκάλεπτη. Και θα μας εξηγήσει πώς αυτή η συμφωνία για διπλή έδρα δημιουργεί προβλήματα στην ε, λειτουργία της ε, υπηρεσίας και θα δούμε και τον κύριο Τίμερ από την Γενική Διεύθυνση Connect για συμπληρωματικά σχόλια. Έχουμε προσκαλέσει και την ελληνική κυβέρνηση για τη συζήτηση αυτή, πρέπει να σας συμπληρώσω, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε ο υπουργό να έρθει μέχρι εδώ. Ο πρεσβευτής που είναι στο Κορεπέρ εκπροσωπείται από τον ε, αντικαταστάτη του, τον καλωσορίζω, τον ε, βοηθό του. Τον καλωσορίζω λοιπόν και θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία οι εκπρόσωποι της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες να μεταφέρουν την πληροφορία και στην Αθήνα, την οποία θα επισκεφθούμε πολύ από εμά στο τέλος του μήνα και πιστεύω ότι θα αποτέλεσε αυτό μια ευκαιρία να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Κύριε Έλμπρεχτ αν έχετε την καλοσύνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα μιλήσω αγγλικά για την παρουσίασή μου. Έχω και κάποιες ε, διαφάνειες ετοιμάσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω μια επισκόπηση της κατάστασης ε, της ενίσας στην Ελλάδα και θα μιλήσω και για την έκθεση απαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εισαγωγικά θα πω ότι θεσπίστηκε το 2004 η ΕΝΙΣΑ με παράταση της εντολής του 2013 έως το 2020 και αξιολόγηση θα γίνει προκαταβολικά για να διατυπωθούν οι προτάσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον κανονισμό του 2013 ελήφθη η μέρημνα και για την έδρα. Αν κοιτάξουμε το ιστορικό, η ένση θεσπίστηκε με αποφάση του Συμβουλίου και ε, Φέθηκε στην κρίση της ελληνικής κυβέρνησης να ορίσει την έδρα το, από το 2003. Αποφασίστηκε λοιπόν το Ηράκλειο της Κρήτης. Το 2013 συμβιβαστικά συμφωνήθηκε οι εργασίες να γίνονται στην Αθήνα και η διοίκηση να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο. Άρα έχουμε περίπου 20 μέλη προσωπικού στο Ηράκλειο και 70 περίπου στην Αθήνα όπω ορίζει ο κανονισμό, Για να κοιτάξουμε λοιπόν τα θέματα που ενδιαφέρουν την ε, ένισα. Ένα από τα κύρια καθήκοντά μας είναι να προσφέρουμε συστάσεις και συμβουλές σε σχέση με την υλοποίηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κοιτάξετε το, την νομοθεσία τη σχετική με την κοινωνία των πληροφοριών, έχουμε τις τηλεπικοινωνίες, ε, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, το κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και άλλους. Έτσι λοιπόν από τα σημαντικά καθήκοντα της ΕΝΙΣΑ είναι να υποστηρίζουν την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στην υλοποίηση του κανονισμού 1S παραδείγματι. Ένα άλλο από τα καθήκοντα της ΕΝΙΣΑ είναι η εξέταση λειτουργικών μοντέλων για την προστασία των δικτύων και τις πληροφορίες και των πληροφοριών μάλλον και να παρέχουν ε, συμβουλές και προειδοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς μπορούν, και τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν να περιορίσουν συνέπειες απειλών, ε, θέματα που έχουν να κάνουν με το cloud computing, το ίντερνετ των πραγμάτων, τα big data, μετρητές ηλεκτρισμού, οικιακούς, υποβοήθηση οδήγηση στα αυτοκίνητα, επικοινωνία μεταξύ αυτοκινήτων και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις απειλές ε, σχετικά με την πληροφορική και την εξυπηρέτηση και των ε, επιχειρήσεων. Έχουμε συζήτηση για την ασφάλεια των ε, πληροφοριών και των δικτύων, όλα αυτά τα θέματα τα οποία υποστηρίζουμε. Και σημαντικός πυλώνας της ε, δουλειάς μας είναι να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Το άρθρο 40, επί παραδείγματι, μας ε, προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν την υποστήριξή μας. Και εμείς αντίστοιχα αναπτύσσουμε ομάδες υποστήριξης. Οι εμπειρογνώμονές μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό, ταξιδεύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, τις Βρυξέλλες, πηγαίνουν σε διασκέψεις κτλ. Και διαχειρίζονται σχέδια. Ο κανονισμός ως προς τη διατύπωσή του συγκεκριμένα. Στην τη σκέψη παριθμών 10 λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσει και περαιτέρω να αναπτύξει τις πρακτικές ρυθμίσεις και την αποτελεσματική λειτουργία. Στη συνέχεια λέει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας κτλ. Σε σχέση με την ισχύουσα τώρα κατάσταση και στην επόμενη διαφάνεια, έχω ετοιμάσει έναν πίνακα Φιρπίν, σε σχέση με την προσβασιμότητα της ε, έδρας τώρα. Έχουμε αμέσες πτήσεις προς το Ηράκλειο για, για και από ε, συγκεκριμένες πρωτεύουσες και μόνο το καλοκαίρι. Γιατί δάλλως οι δραστηριότητες στο Ηράκλειο είναι είτε γεωργικές είτε τουριστικές. Άμεσες πτήσεις λοιπόν έχουμε από την Αθήνα μόνο προς τους κύριους ευρωπαϊκούς προορισμούς σε, στη διάρκεια ολοκληρού του έτους σε σχέση με τις δυνατότητες τις εκπαιδευτικές, ε, τα σχολεία. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχολείο στο Ηράκλειο. Δυστυχώς όμως η πρόκληση μεγάλη είναι ότι δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα μαθητών ώστε να προσφέρονται όλες οι τάξεις. Η μεγάλη μας πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει σωστά λειτουργούσα δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έκθεση της ε, αξιολόγησης για τα ευρωπαϊκά σχολεία που αφορά το Ηράκλειο ε, οδηγεί σε σπεράσματα ανησυχητικά γιατί φαίνεται να μην εξασφαλίζει στο μέλλον την πιστοποίηση ως ευρωπαϊκό το σχολείο αυτό του Ηρακλείου. Για την Αθήνα τώρα έχουμε πολλά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και σε επίπεδο διεθνών ε, σχολείων έχουμε γερμανικά, αμερικανικά, γαλλικά Άρα μεγάλο φάσμα επιλογών για τους γονείς, για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στο τρίτο κομμάτι αυτού του πίνακα, πρόσβαση προς την αγορά εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθεψη για παιδιά και συζύγους. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που όπως είπα δεν είναι σύστημα, οικοσύστημα καλύτερα πληροφορικής ή ασφάλειας των δικτύων. Όπως είπα, ως περιοχή έχει περισσότερο γεωργία και τουρισμό. Οι σύζυγοι επιτοπλίστων δεν μπορούν να βρουν ε, δουλειά. Πολλές φορές ε, οι υπάλληλοι μας χρειάζεται να ταξιδεύουν, να ταξιδεύουν ε, και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης ακόμη τα Σαββατοκύριακα και αυτό σημαίνει πολύ σημαντική επιβάρυνση. Άρα είναι δύσκολο να βρούμε, να προσελκύσουμε ε, αρκετούς ενδιαφερομένους για να εργαστούν εκεί. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την ε, έκθεση απαλλαγής του 2013 με τις δύο αυτές έδρες ρητά αναφερόμενες και το σχόλιο εδώ είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επίσης ε, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα αυτής της διπλής έδρας. Πολλές συζητήσεις λοιπόν και και στην έκθεση απαλλαγής καταγράφεται ότι και το κόστος από την ενοικίαση είναι σημαντικό. Αν δούμε την κατάσταση στο, στα κτίρια της Αθήνας, το ενίκιο το καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση και αισθανόμαστε ευγνώμονε γι' αυτό γιατί πρόκειται για σημαντικό ποσό. Αλλά η πρόκληση είναι ότι ο ε, εκμισθωτής, ο ιδιοκτήτης ε, πληρώνεται μόνο τελευταία στιγμή και πολλές φορές με αρκετές δυσκολίες. Μπορούμε εμείς να παρέμβουμε για να φτάσουν στα χέρια του τα χρήματα. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα ο ε, ιδιοκτήτης έχει δείξει πολύ καλή διάθεση, έχουμε ωραία γραφεία κτλ. Αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην πληρωθεί εγκαίρως στο μέλλον το νίκη. Τώρα πρακτικά τι συνέπειες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι συμβιβαστικά ο κανονισμός, πολιτικός συμβασμός δηλαδή ήταν, ε, και όριζε την διοίκηση στο Ηράκλειο και τη λειτουργία στην Αθήνα. Ύστερα από αυτά τα τρία χρόνια περίπου βλέπουμε να μην λειτουργεί αυτό το σύστημα, παραδείγματι. Στην πληροφορική χρειάζεται προσωπικό που θα έχει έναν υπολογιστή που θα λειτουργεί σωστά μέσα στο γραφείο του. Δεν μπορεί να ταξιδεύει ο υπάλληλο από το Ηράκλειο στην Αθήνα αν έχει κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή του και άρα η δουλειά αυτή της πληροφορικής μοιράζεται ανάμεσα στην Αθήνα και το Ηράκλειο. Εάν υπάρχουν θέματα ανθρωπίνων πόρων, ε, συνεντεύξεις για κάποιο νέο υποψήφιο, θα πρέπει να πάει κανείς στην Αθήνα για να του συναντήσει και Τούμπαλιν ε, για τις ε, προμήθειες, το γραφείο των προμηθειών στο Ηράκλειο, ενώ το έργο μπορεί να το διαχειρίζεται το Αρφείο των Αθηνών, οπότε πρέπει να μεταβούμε στην Αθήνα. Πολλές, ε, πολλά είναι τα, σημεία και τα προβλήματα που είναι αποτελεσματικότητα. Στα δεξιά μου, ο Πάλλο Παντένια που είναι επικεφαλής της διοίκησης έχει ε, ως προς τα ηλεκτρονικά μέσα καταφέρει πολύ σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο πολλά πράγματα ακόμα ε, συνεπάγονται ταξίδι για τους υπαλλήλους μας για να μην αναφέρω εκείνους που φεύγουν σε αποστολή και πρέπει να περάσουν από το Ηράκλειο στην Αθήνα για να μεταβούν σε μια άλλη πόλη της Ευρώπης, άρα χάνουν πολύ χρόνο όσοι ταξιδεύουν. Άρα το κόστος της, αποστολής μας, της επιτέλεσης αποστολής μας ε, γίνεται πιο υψηλό. Έχουμε πρόβλημα προς την επικοινωνία. Στην πρακτική, αν υπάρχουν δύο έδρες, είναι δύσκολη και η επικοινωνία μεταξύ των μελών του προσωπικού, ναι, οι υπάλληλοι μπορεί να μην γνωρίζονται καν με τους άλλους και τελικά η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου είναι πολύ ε, λεπτή και είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουμε σε αυτή την ε, αγορά σε αυτό, ε, νέο προσωπικό, γιατί πάντα έρχεται κάποιος να μου πει «Μα τι θα κάνω τώρα, τόσο με το σχολείο των παιδιών μου που μεγαλώσαν, πρέπει να πάω στην Αθήνα για να δουλεύω από εκεί, γιατί εκεί μπορούν να έχουν καλύτερες ευκαιρίες για σχολείο τα παιδιά μου». Όλα αυτά μαζί νομίζω τα δείχνουν πολύ ικανοποιητικά δύο αριθμητικά στοιχεία. Για να σας πω το εξής με μία μονοέδρα και αυτό αποτελεί μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξοικονομούσε το 40% από το κόστος του ενοικίου. 40% εξοικονόμηση από το κόστος του ενοικίου για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί εκείνη καταβάλει τα ενίκια. Για μας η επιβάρυνση λειτουργική θα μειωνόταν κατά 6% από τον προπολογισμό που τώρα χάνουμε ως προς την αποτελεσματικότητα και θα μπορούσαμε να διαθέσουμε σε έργα και project με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε την ε, παραγωγή μας. Έτσι λοιπόν η τωρινή εντολή όπως είπα πάει μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Έχουμε μια αξιολόγηση που ξεκίνησε η Ενίζα πέρυσι και θα συνεχιστεί και φέτος για να προετοιμάσουμε την αξιολόγηση. Βέβαια η αποτελεσματικότητα και τα σημεία που ανέφερα εδώ επίσης θα καταγράφονται στην έκθεσή μας και με το βλέμμα προς το μέλλον νομίζω πρέπει να συζητηθεί και να συζητήσουμε το μέλλον της εντολής. Χρειάζεται μια αποτελεσματική υπηρεσία που θα καλύπτει τις ανάγκες στην ασφάλεια των δικτύων και της ε, πληροφορίας και γι' αυτό θέλουμε να μας υποστηρίξετε ώστε η ενίσχυση στο τέλος να ε, έχει μόνο μία έδρα και εν προκειμένου την Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τίμερς είναι ο επόμενος ομιλητής. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και για να πω δύο λόγια στα γρήγορα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, το θέμα αυτό, γιατί η Γενική Διεύθυνση Connect βεβαίως παρακολουθεί ε, πολύ στενά τις δραστηριότητες της ΕΝΙΖΑ και βέβαια και κάθε εξέλιξη σε ε, επίπεδο χάραξης πολιτικής. Το 2004 ο καθηγητής μας το εξήγησε πολύ καλά όταν ιδρύθηκε αυτή η υπηρεσία η απόφαση ελήφθη να εγκατασταθεί στην Ελλάδα και υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη. Κατόπιν στον κανονισμό του 2013 που καταργούσε τον προηγούμενο κανονισμό και που ε, ψηφίστηκε και από εμάς και από τα κράτη-μέλη, αναφέρθηκε πως για λειτουργικούς ε, λόγους και για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ε, θα εγκατασταθεί και ένα τμήμα αυτή στην Αθήνα. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα είναι η γραμμή που με απασχολεί και εσείς ως ε, Επιτροπή ε, στα σχόλιά σας ε, κατά την διαδικασία απαλλαγή είναι πολύ σημαντικό η στρατηγική λειτουργικότητα να αυξηθεί γιατί έχουμε πάρα πάρα πολλέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στον κυβερνοχώρο. Διαβάζετε τι συμβαίνει στι εφημερίδε και για τη χάραξη πολιτικής και την εξέλιξη των πολιτικών μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πάρα πολλά. Έχουν αποφασιστεί πολλά και από εδώ και από τα κράτη-μέλη. Έχουμε την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων, για παράδειγμα, και των πληροφοριών, όπου έχουμε στρατηγική και ε, λειτουργική ε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στην οποία συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό και η ΕΝΙΖΑ. Ένας από τους κανόνες ε, στην ΕΝΙΖΑ είναι ε, για την κυβερνοασφάλεια να είμαστε κομβικό σημείο για ολόκληρη την Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε βέβαια πως η ΕΝΙΖΑ αντιμετωπίζει θέματα που σχετίζονται με την καταβολή του μισθείου για τα δύο γραφεία, όπου η ελληνική κυβέρνηση με πολύ γενναιόδρο και ευγενικό τρόπο ε, προσφέρει τη στήριξή της και σε αρκετές περιπτώσεις ήρθαμε σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε κατόπιν αιτήματος της ΕΝΙΖΑ πώς θα καταβάλλεται πρόθεσμα το μισθείο, αλλά το να καλύπτονται τα έξοδα αυτά της ΕΝΙΖΑ είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης και παραμένει θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν επιχειρησιακές και λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υπηρεσία με τα δύο αυτά ξεχωριστά γραφεία και είμαστε πολύ συχνά σε επαφή και με τον διευθυντή και με την ίδια την υπηρεσία για να δούμε ποιος είναι ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της τρέχουσας κατάστασης. Προβλέπεται από τον κανονισμό του 13 στο άρθρο 32 να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα ε, της ΕΝΙΣΑ τον Ιούνιο του 2018 έτσι ώστε να έχουμε μία εντολή, μία ανανέωση εντολής της ΕΝΙΣΑ ε, που θα λαμβάνει υπόψη ε, το πώς θα έχει τρέξει κατάσταση με την ε, αποτελεσματικότητα, τη λειτουργικότητα αλλά και με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Όλα αυτά λοιπόν θα ληφθούν, θα ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από τον κύριο Γκαγέ, Γκάγερ που είναι ο μόνιμος εισηγητής για τα θέματα αυτά να μας πει και αυτός δύο λόγια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είναι άγνωστο το πρόβλημα αυτό στην Ευρώπη. Έχουμε και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες που έχουν διαφορετικές έδρες και όλα αυτά προκύπτουν κατόπιν πολιτικών αποφάσεων. Κάποιες από αυτές μπορούμε να τις ανατρέψουμε και άλλες όχι. Και έτσι τίθεται το ερώτημα. Ε, οι υπηρεσίες που έχουν δύο έδρες μπορούν να αλλάξουν καταρχάς έδρα, αλλά όχι με δική μας απόφαση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ε, υπάρχει καμία δυνατότητα. Ξέρω καλά την περίπτωση της Ενίζας, την τελευταία θητεία και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχα παρακολουθεί στην υπόθεση με την απαλλαγή και τις εκτιμήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Τα γνωρίζω όλα αυτά πολύ καλά και ο Γενικός Διευθυντής πολύ σωστά τα περιέγραψε. Κύριος Χέλμπρεχτ. Είναι γνωστό ότι όταν υπάρχουν διπλές έδρες τα πάντα περιπλέκονται και όταν χρειάζεται να πάρει κανείς το φεριμπότι το αεροπλάνο για να πάει από τη μία ε, πόλη στην άλλη, από τη μία έδρα στην άλλη, ακόμα περισσότερο βάλιστα. Είναι δύσκολο να βρεθεί το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για τη δουλειά της ΕΝΙΖΑ. Υπό τις συνθήκες εκείνες ε, βεβαίως ήδη με τον πολιτικό συμβασμό, αλλά ήδη μας περιέγραψε ο κ. Σέλπρεχτ τα προβλήματα, άρα και ως προς την αποτελεσματικότητα και ως προς την εξοικονόμηση πόρων θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενοποιήσουμε τις δύο έδρες της ΕΝΙΖΑ. Και αν πρόκειται για πολιτική απόφαση και αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση έστω να πάρει τη σχετική απόφαση. Αλλά ο κανόνα ισχύει και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κάθε χώρα που υποδέχεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, ότι τη λειτουργία της υπηρεσίας την εξασφαλίζει η κυβέρνηση, η χώρα υποδοχής. Και εδώ το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ το ποσό στο οποίο συμμετέχει ο καθένα, τόσο ή άλλω είναι γνωστέ οι δυσκολίε οικονομικέ τη ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ίσω αν και δυσανάλογη δηλαδή η επιβάρυνση, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία Μα ε, ανησυχούν και γι' αυτό απευθύνω κατεπίγουσα έκκληση προ την ελληνική δημοκρατία, προ το ελληνικό κράτο, να ξαναεξετάσουν αυτά τα ζητήματα και να επιτρέψει στην Ενίζα με όλο της το προσωπικό να μεταφερθεί στην Αθήνα ή μη τι άλλο σε, μια τοποθεσία πολύ πιο προσβάσιμη από το Ηράκλειο της Κρήτης. ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα σημείο, να επικεντρώσει σε ένα σημείο. Ανέφερε και ο Γενικός Διευθυντής ότι θα επανεξεταστεί η εντολή της υπηρεσίας του 2020. Επομένως, τουλάχιστον μέχρι τότε θα μας, τουλάχιστον τότε θα μας, επανεξε, θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα της υπηρεσίας. Βέβαια, μέχρι τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει κάποια συμπεράσματα για τη δουλειά της ΕΝΙΖΑ και είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εγκρίνει για άλλη μια φορά κατάσταση κατά την οποία μια υπηρεσία είναι κατανεμημένη, έχει κατανεμημένες έδρες σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Εγώ Πιστεύω ότι το 2020, τη στιγμή που θα πρέπει να ε, γίνει η επεξεργασία του νέου κανονισμού, θα είμαι ακόμη ευρωβουλευτής προκειμένου να με ρημνήσω ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό απευθύνω προς τις κυβερνητικές αρχές, προς τις κρατικές αρχές Ελλάδας, να μην αφήσει το πράγμα να χρονίσει μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Εισηγητή μας και ελπίζω οι ελληνικές αρχές να εισάκουσαν την έκκλησή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Στεχόφσκι. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Τι νόημα έχει αυτή η παρουσίαση. Γιατί εγώ ελπίζα να καταλάβω γιατί να έχει δύο έδρες αυτή η υπηρεσία. Όμως το μόνο που άκουσα ήταν περισσότερα επιχειρήματα για το πώς πρέπει να απαλλαγεί από τη μία από τις δύο έδρες η υπηρεσία. Γιατί έχει δίκιο ο κύριος Γκάιερ. Είναι πολλά αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουν. Οπότε ή θα πρέπει να καταργήσουμε τη δεύτερη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο, αύριο ή και την τρίτη έδρα στο Στασβούργο και στο Λουξεμβούργο αντίστοιχα. Γιατί εν προκειμένου νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ζήτηση που να στέκει. Να μιλήσουμε για την αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας η οποία ε, έχει τις δύο έδρες και συμφωνώ με όλα όσα αναφέρθηκαν γιατί μίλησα με κάποιους που είπαν ότι ποτέ δεν πρόκειται να πάνε εκεί να υπηρετήσουν ποτέ δεν θα ήθελαν να μένανε εκεί υπάρχει πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Σχολείο το οποίο δεν μπορεί να αποσπάσει μια επιστοπίσμα τι άλλα επιχειρήματα χρειάζονται Καμιά φορά θα πρέπει κανείς να αποδεχθεί ότι μια υπόθεση απέτυχε. Και εμείς που εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν συντρέχουν τέτοια περιστατικά κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Να, τι πάει στραβά σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως ε, σε κάποιους δεν αρέσει το τι στο παίρνω, αλλά οι περισσότεροι δυσαρεστούνται από το πώς διασπαθίζουμε, πώς, πού, πού, πού πάνε τα χρήματα των φορολογουμένων, τι θα κάνουμε. Και έριξα μια ματιά στα σχετικά με την υπηρεσία αυτή, η Κρήτη είναι υπέροχο νησί, λατρεύω την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι υπέροχη τόπη. Από πλευράς τώρα του να δαπανάει και τους κοινωτικούς πόρους για να συντηρεί μια υπηρεσία χωρισμένη σε δύο έδρες, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι φύρα, είναι απόλυτη αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει προκειμένου να μιλήσουμε για το Brexit. Μα πώς να πιστεί κανείς ότι είναι αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δει τι γίνεται με αυτή την υπηρεσία. Γιατί Υπάρχουν τέτοια προβλήματα και για άλλες υπηρεσίες. Ελπίζω ότι θα παραμείνει η υπηρεσία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί η Ελλάδα για να βοηθήσει την υπηρεσία. Αλλά τι να συζητάμε για έδρα της ε, ε, υπηρεσίας. Δεν ζητεί άλλο το λόγο λέει ο πρόεδρος. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος. Και να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο που τον ζήτησε. Ναι, συμφώνω, ε, συμφώνω ότι και σαν Επιτροπή Προπολογισμών εμείς πάντοτε θα πρέπει να επιδιώκουμε εξοικονομίζει δαπανών. Και εγώ ίδιο συμφωνώ. Ναι, ναι, λέει ο κύριος ε, Κίρτσο, συμφωνώ με αυτή την επιχειρηματολογία. Ε, νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά τα είπαν οι πρόσωποι της υπηρεσίας, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία μόνο έδρα, μάλλον στην Αθήνα. Και έχω ε, κάποια καλά μαντάτα για σας παρά το ότι προέρχομαι από το κόμμα της εξωματικής στην Ελλάδα. Νομίζω η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να συνεργαστεί. Βέβαια πρόκειται να αναφύγουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ντόπια πολιτική. Αλλά βέβαια είναι κατανοητά τα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ελλάδα και θα εξευρεθεί αναγκαία λύση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το θέμα. Άρα λοιπόν θα θέλαμε η κατάσταση αυτή να ξεπεραστεί έτσι ώστε να μην βλάβεται η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών, να μην γίνεται κατασπατάληση πόρων και εμείς, όπως πρότεινε ο μόνιμος συγητής μας, είπαμε πως θα προτείνουμε να λήξει αυτή η κατάσταση. Εγώ θα είμαι στην Αθήνα τέλη του μήνα και θα μιλήσω με τον αρμόδιο υπουργό για να μου επιβεβαιώσει πως η κατάσταση αυτή, η αφύσικη αυτή κατάσταση θα λήξει. Ας το αφήσουμε λοιπόν εκεί και να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι τα ομόλογα έργου. Δυστυχώς ε, σε μισή ώρα εγώ πρέπει να φύγω αλλά έχουμε εδώ τον συνάδελφο ο οποίος θα αναλάβει ε, το, την Προεδρία, τον κύριο Σαραβαμά. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 11 της μυρίσιας Θα είναι τα ομόλογα έργου. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Νίκ Τζένετ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας σήμερα εδώ. Είναι η πέμπτη ε, φορά που συναντιόμαστε για τη μηνιαία έκθεση πεπραγμένων και βεβαίως τώρα που προχωράμε προς το τέλος της πιλωτικής φάσης τα πράγματα επιταχύνονται. Ως εισαγωγή να σας υπενθυμίσω πως η πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 με στόχο να αναζωπυρώσουν την χρηματοδότηση των κερδοσκοπικών αγορών, κυρίως στο θέμα των υποδομών και κυρίως στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και δίκτυα ενέργειας. Και βέβαια, η ανάγκη αυτή προέκυψε Αν κοιτάξετε το διάγραμμα επάνω δεξιά στη γωνία, που αναφέρεται ότι πριν την χρηματοστητική κρίση οι αγορές ήταν αυτές οι οποίες επενδύανε στις υποδομές στην Ευρώπη. Ήταν δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, τα μία ταμεία τα οποία ε, χρηματοδοτούσαν ε, τις μακροπρόθεσμες υποδομές στην Ευρώπη με την έκδοση ε, ομολόγων για έργα τα οποία ε, εκτελούσαν μεγάλες εταιρείες. Με την χρηματοπιστική κρίση δυστυχώς αυτό το είδος χρηματοδότησης έληξε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Project Bond Initiative με σκοπό να συνδυάσουμε τους πόρους που έχει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός και η ΕΤΕ έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε project υψηλής αξίας σε όλη την Ευρώπη αλλά επίσης για να αναπτύξουμε και ένα καινούριο τρόπο χρηματοδότησης όπου ε, αυτά τα ομόλογα έργο ένας τρόπος χρηματοδότησης αυτών των τόσο πολυδάπανων project. Από τότε που ξεκινήσαμε, 9 και πολύ σύντομα 10 project έφτασαν μέχρι τις αγορές με τη συμβολή αυτών που έχουμε τον PBCE, έτσι το ονομάζουμε εμείς, που είναι το Project Bond Credit Enhancement, αν δείτε πάνω δεξιά στην ε, διαφάνεια ε, και κοιτάξτε εκεί το διάγραμμα, θα δείτε πως όντως ε, πραγματικά επηρέασαν, γιατί από το 2012 το ποσοστό των υποδομών σε όλη την Ευρώπη καινούριων υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από τις έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Η πρωτοβουλία αυτή στόχευσε σε τρεις χώρους πολιτικής προτεραιότητας. Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορές, ενέργεια και ευρυζωνικότητα. Και ουσιαστική εταιρική σχέση μεταξύ τραπεζών και ε, ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ήταν τα 230 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατέθησαν στην τράπεζά μας καταρχήν ως ε, αρχικά κεφάλαια σε χαρτοφυλάκια για επενδύσεις σε αυτούς τους τρεις κλάδους σε περιπτώσεις όπου η ΕΤΕ χρησιμοποίησε τη στήριξη και τις πιστώσεις αυτές από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τα 230 εκατομμύρια, έτσι ώστε να εκδώσει και χρηματοδοτούμενα και μη χρηματοδοτούμενα ε, ε, τέτοια PBCE έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως τα ομόλογα που οι διάφορες εταιρείες εξέδιδαν θα είχαν αρκετή, ε, ε, ε, θα ήταν τέτοιες βαθμολογίες που θα ήταν ελκυστικά για, τις, για τα ασφαλιστικά ταμεία και τα εξαιρετικά ταμεία ως επενδυτική δυνατότητα. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στο να μπορούμε να στηρίξουμε γύρω στα 3,5 δις ευρώ δανείων και δαπανών, σχεδόν 4 δις ευρώ, μόχλευση δηλαδή της τάξης, ε, ε, ενός πολλαπλασιαστή της τάξης του 19 φορές ε, παραπάνω από το αρχικό ε, κεφάλαιο που ήταν διαθέσιμο. Αυτά βεβαίως χρειάστηκε και μέχρι το 2014 να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ. Άρα λοιπόν το χαρτοφυλάκιο έχει πλέον οριστεί και έχουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 έτσι ώστε τα project αυτά σε χρηματοδοτικό επίπεδο να έχουν κλείσει. Να πω και δύο λόγια γρήγορα για τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά λειτουργούν. Η ΕΤΕ εκδίδει τέτοιου είδους ε, δάνεια, είτε χρηματοδοτη... δευτερεύοντα ε, ε, δάνεια, τα οποία είτε έχουν χρηματοδοτηθεί από την ίδια τη τράπεζα, είτε από κάποιους δανειστές, είτε εκδίδει μερικές εγγυήσεις ως δευτερογενή δάνεια και οι χρηματοδοτούμενοι και οι μη χρηματοδοτούμενοι μορφή μπορούν να φτάσουν και το 20% του συνολικού ομολόγου έργου που μας οδηγεί σε ένα credit enhancement που είναι παραπάνω από τα μετοχικά κεφάλαια τα οποία έχουν σημειωθεί για τα ομόλογα αυτά, το οποίο σημαίνει ότι οι εταιρείε μπορούν να εκδώσουν ε, συν τρία σε σχέση με την αρχική τους βαθμολογία, δηλαδή μπορούν να φτάσουν και στο A- ως αξιολόγηση για τα ομόλογα αυτά τα οποία εκδίδουν. As of today, some six... Έχουμε έξι τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει μέχρι σήμερα έξι τέτοια εγχειρήματα με στήριξη του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού σε πέντε κράτη-μέλη και θα δείτε εδώ στη σελίδα ποια είναι ε, αυτά. Έχουμε μεταφορές, ευρυζωνικότητα και τις σχετικές υποδομές και ενέργεια. Με project διαδίκτυα ε, στις μεταφορές καλύπτουμε την γάμα μεταξύ οδικών αξώνων, ε, δηλαδή έχουμε και ε, αυτοκινητοδρόμους και λιμάνια και επιπλέον λόγω των περιορισμών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκά κονδύλια προς τη στήριξη αυτών και επειδή είχαμε θύματα από όσους προτείνανε έργα έχουμε κλείσει και δύο project σε δύο κρατημέλη χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αν έχουμε λοιπόν, αν δείτε αυτές τις, ε, τα εννέα εγχειρήματα, έξι στηρίζονται και τα υπόλοιπα βρίσκονται μόνο στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, θα δείτε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν τα 6 δις ευρώ 4,5 δις έχουν εκδοθεί ως ομόλογα έργο και όλα αυτά με κάλυψη ε, PBCE της τάξης του 0,7 δις. Θα κάνω λοιπόν εδώ μία σύνοψη για τα project τα οποία έχουν στηριχθεί και θα σας πω πως αυτά που πετύχαμε είναι αυτά τα οποία σας παρουσίασα και αν συμφωνείτε κι εσείς θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο, στον Τζόρτζιο Κασόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σας εξηγήσει πώς έχει αξιολογήσει τις επιδόσεις μας μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Είναι η πέμπτη φορά αυτή που παρουσιάζουμε τη συμβολή μας ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τα ομόλογα, για των έργων και έχουμε αυτήν την ε, νομική βάση και κάνουμε αυτή την εξωτερική αξιολόγηση για την ε, πρωτοβουλία ομολόγων έργων και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση τον Δεκέμβριο του 2015. Και ακριβώς αυτά και σας αναφέρουμε σήμερα. Αυτή η αξιολόγηση έλαβε υπόψη την προσθετικότητα της ε, πρωτοβουλία των αιμορροπινών σε σχέση με άλλα μέσα. Και η επίπτωση αυτής της φάσης, όπως ε, προαναφέρθηκε, ε, ξεκίνησε χρονικά από τη στιγμή που η χρηματοδότηση του χρέους ήταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οπότε και υπήρξε ένα άλλο μέτρο που θέλαμε να αξιολογήσουμε τον πολλαπλασιαστή σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και να αναλύσουμε την ανταγωνιστικότητα της λύσης των ομόλογων έργων σε σχέση με άλλου είδους ε, εργαλεία ή μέσα. Για να δούμε τώρα το χρονικό πλαίσιο, μιλάμε τον Ιούλιο του 2015 και να μην επαναλάβω τα στατιστικά στοιχεία απλώς να σας αναφέρω ότι ο αρχικός στόχος ήταν να έχουμε 7 έως 10 κινήσεις σε αυτή την πιλωτική φάση. Τελικά δηλαδή, είχαμε 10 τέτοιες κινήσεις που ε, καλύφθηκαν από τον προϋπολογισμό μας και 7 από τον κοινωτικό προπολογισμό. Και έγινε με τι συνήθειε διαδικασίε η αξιολόγηση. Επίση, κάναμε διάφορε συνεντεύξει με του εξωτερικού εμπλεκόμενου. Είχαμε επομένω 7 προγράμματα ή έργα τα οποία αξιολογήθηκαν ε, μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Αλλά τρία ε, έργα τα οποία έχουν γραμματωθεί μέχρι τώρα και θα συμφωνηθεί ακόμα ένα έργο τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αν μπορεί να έχει να απαντήσουμε. Τώρα, όσον αφορά μια σύνοψη των συμπερασμάτων μας, των διαπιστώσεων, ας πούμε, το σημαντικό είναι το ότι από πλευράς αποτελεσματικότητας, το πιο σημαντικό στοιχείο που βγήκε από αυτή την πιλωτική φάση είναι ότι η αγορά των έργων ε, ήταν σε νεκρό σημείο και για τις ε, εξατομικευμένες δράσεις αλλά και για τις κοινέ ε, της ε, ΕΤΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθειες δηλαδή για να αναζωογονηθεί η αγορά. Οπότε είχαμε αυτή την πρωτοβουλία των ομολογών έργων και αυτό αναζωογόνησε κάπως την αγορά. Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε πιο πολλούς θεσμικούς ε, επενδυτές σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από λίγα χρόνια. Και οπότε ε, έχουμε επομένω και από πολιτική πλευράς υποστήριξη της προσπάθειας. Είπαμε για διαφορετικού κλάδου, διαφορετικά μέρη και αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε από αυτή την πρωτοβουλία αν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε κάπου αλλού, κάποια άλλη στιγμή την εφαρμογή αλλίου. Οπότε οι θεσμικοί επενδυτές έτσι δεν τη θέση τους να ενισχύεται και είδαμε να υποστηρίζει καλύτερη χρηματοδότηση. Όλα αυτά τα έργα είπαμε ότι είναι επιλέξιμα, θεωρούνται έργα πρωτοβουλίες και η ιδέα μόχλευση όπως τα σας τα εξήγησε ο Νίκ μας οδήγησε στο να πετύχουν, όπως λένε και τα στατιστικά στοιχεία, να πετύχουμε σε αυτά τα επτά έργα του κοινωτικού προϋπολογισμού. 19 ε, ε, φορές ε, ήταν ο πολλαπλασιαστής και το, ε, η μόχλευση. Και πήγαμε στα 230 εκατομμύρια όσον αφορά τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό. Τώρα ανακλάδω όπως και περιμέναμε, ήταν αλλιώ τα πράγματα σε κάθε αγορά, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αυτά τα ομόλογα έργων ε, απεδείχθησαν ότι ήταν το, το πιο δόκιμο μέσο όσον αφορά τον κλάδο της ε, ενέργειας, ιδίως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένο εργαλείο ε, και η ΕΤΕ επίσης συνέχισε την χρηματοδότηση, επίσης τα, τα ευρωζωνικά και εκεί τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν το μόνο έργο που έγινε σε αυτόν τον κλάδο στην ε, Ευρώπη. Οπότε φάνηκε ότι έτσι μπορούμε να κάνουμε και άλλα τέτοια έργα για τα ευρωζωνικά με τον ίδιο τρόπο. Τα πιο μεγάλα και τα πιο μικρά που πολλές φορές αποκλείονται. Και το όφελος ήταν ότι έτσι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια έργα Greenfield γιατί θα πρέπει να καλυφθούν στην πιλωτική φάση οι κίνδυνοι που προκύπτουν. Και έχουμε καλύτερα μακροπρόθεσμα έργα και όσον αφορά τις δαπάνες κεφαλαίου και όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Αλλά θα πρέπει να πετύχουμε και καλύτερες τιμές, κάτι το οποίο έχει σημασία για τον δημόσιο τομέα που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό κατακύρωσης του έργου. Οπότε από τις ε, συνεντεύξεις φάνηκε ότι η συμμετοχή της ΕΤΕ και στον διαγωνισμό και μετά ε, ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό που εκτιμήθηκε και ε, βοήθησε στο να δείξει ότι θα ολοκληρωθεί το έργο γιατί ακριβώς ένιωσαν καλά, πολύ, πολύ θετικά οι επενδυτές ότι συμμετέχει η ΕΤΕ και ότι θα του συνοδεύσει σε όλη αυτή την πορεία του έργου. Σε όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις που μελετούμε φάνηκε αυτό και στις αξιολογήσεις μιλάμε για δύο-τρία κλικ κάθε φορά που προέκυψαν από τη στιγμή που υπήρξε η ανακοίνωση του ομόλογου έργου. Τώρα όσον αφορά την επίδειξη των στόχων της πολιτικής, να μην επαναλάβω, ήταν κάτι σημαντικό στην πολιτική φάση και στην αξιολόγηση προέκυψε ότι αλλάζει η αγορά, τώρα υπάρχει περισσότερη ρευστότητα. Και χάρη σε αυτό το εργαλείο και χάρη στην ε, ε, Ένωση της Κεφάλαια Αγοράς και από τις τράπεζες και από τους θεσμικούς ε, επενδυτές ε, οι οποίοι προσήλθαν για να συμμετάσχουν άρα στο μέλλον θα πρέπει λέει η αξιολόγηση να αρθούν κάποια πάρα πολύ κενά που υπάρχουν ε, στις υποδομές της να συνεχίσουμε να έχουμε έργα Greenfield και επίσης να προσέξουμε γεωγραφικά που γίνονται αυτά και σε ποιον κλάδο. Ε, επίσης είπαμε ότι το εργαλείο έχει πολύ καλά σχεδιαστεί και βεβαίως ε, η εμπειρία μας έμαθε κάποια πράγματα, το πώς λέει θα προσαρμοστεί το έργο και κατά πόσο ανάλογα με το έργο πώς υποστηθέμενη αξία υπήρχε ας πούμε σε κάποια έργα για τις μεταφορές όπου η ανακοίνωση, η προκήρυξη των ομολόγων προσαρμόστηκε ε, στην εξέλιξη του έργου και δεν εκδόθηκαν τα ομόλογα όλα μαζί. Και ε, τώρα λοιπόν που η αγορά έχει πιο πολύ ρευστότητα, έτσι θα συνεχίσουμε και θα επικεντρωθούμε στους κλάδους εκεί που η αγορά τα πάει χειρότερα. Ωρα. Σαν συστάσεις μπορούμε να πούμε ότι η αξιολόγηση έδειξε ότι αυτό το προϊόν το χρειάζεται η αγορά και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Τραπέζα Επενδύσεων θα πρέπει να να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν για τα έργα υποδομής θα πρέπει να συνεχιστεί η μόχλευση από τον κοινωτικό προϋπολογισμό να μην σταματήσει η ΕΤΕ συμμετοχή της έτσι δεν θα αποκτήσει γνώση, εμπειρία η αγορά, αλλά αυτό θα είναι και ένα αρνητικό μήνυμα προς τις κεφαλαίες αγορές και τους επενδυτές στα έργα υποδομής. Εάν σταματήσει την υποστήριξη ή είτε γιατί αυτό θα αντιβαίνει στο πνεύμα της Ένωση κεφαλαίων Επίση, για την αποτελεσματικότητα αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να εστιαστούμε περισσότερο σε κάποιου κλάδου, σε κάποια μέρη όπου υπάρχει και κοινωτική προστεμένη αξία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι με παρόμοιο πνεύμα και η ε, Ένωση και η ΕΤΕ προχώρησαν σε αυτό το όργανο για να διευρυνθεί αυτό το φάσμα των προϊόντων και να μην είναι περιορισμένος ο ορίζοντας των οργάνων που χρησιμοποιούμε. Γιατί θέλουμε να έχουμε και στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στην ενέργεια, κάποια διασυνοριακά ε, εργαλεία και να υπάρχει και εταιρική χρηματοδότηση ανάλογα με αυτό το οποίο χρειάζεται κάθε φορά και το τι είναι η πιο αποτελεσματική λύση. Αλλά μοιάζουν οι δομές αυτής της ε, πρωτοβουλίας Οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια και να κάνουμε τα ίδια και ε, στο Connecting Europe Facility. Να καλύψουμε νέους κλάδους, χώρες, έργα και είναι σημαντικό να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν όχι μόνο από το Connecting Europe Facility αλλά και ε, το καινούριο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και σε κάποιους τομείς όπου υπάρχει έντονο ενδιαφέρον το να υπάρξουν ε, ομόλογα έργο, οικονομία, ε, μειωμένο άνθρακα, σε αυτούς τους, σε αυτούς τους κλάδους, σε αυτούς τους τομείς πυρήνες. Οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε με αυτή τη θετική αξιολόγηση τι θα γίνει με αυτό το προϊόν ε, για το Connecting Euro Facility, γιατί είπαμε ότι το 2016 ολοκληρώνει την πιλωτική φάση για τα ομόλογα έργο. Οπότε τότε δεν θα είναι κάτι το ξεχωριστό σαν πρωτοβουλία, αλλά θα έρθει να ενωθεί με τις προηγούμενες πρωτοβουλίες του Connecting Euro Facility, την πρωτοβουλία σχετική με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, Οπότε η χρήση των ομολόγων δεν θα περιοριστεί εκεί, θα είναι ακόμα ένα προϊόν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή του Ταμείου Στατικικών Επενδύσεων ή του Γενικού Παιδικού Πλάνου για την Ευρώπη και επομένως είναι σημαντικό για να τα πάμε καλά και η Τράπεζα Επενδύσεων να χρησιμοποιήσει όλες τις ε, δυνατότητες ούτως ώστε να ενημερωθούν όσο γίνεται περισσότεροι και βέβαια να υπάρχει εξειδικευμένη γνώση για αυτή την δραστηριότητα. Θα συνεχίσουμε επομένω να εξετάζουμε το πού δεν τα πάει καλά η αγορά, ιδίω για τα διασυνοριακά έργα και για τις ε, λιγότερο ενεργές αγορές. Όλα αυτά για τις υποδομές στην Ευρώπη. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο λοιπόν. Ο εισηγητής για το θέμα αυτό είναι η κυρία Έτσια. Πάλι δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά κάνατε μια πολύ καλή παρουσίαση του πώς λειτουργεί ε, το θέμα αυτό των ομολόγων έργου και κυρίως για την πιλωτική φάση. Και με τις συνόψεις που μας κάνατε νομίζω πως η πρώτη αυτή φάση ήταν πολύ ικανοποιητική. Κάτι το οποίο δεν έχω καταλάβει είναι τι συνέχεια θα δώσουμε αφού ξεπεράσουμε ε, την ε, πιλωτική φάση. Δηλαδή, ε, με το πακέτο Juncker και με το Connecting Europe θα συνεχίσουμε ή ε, θα σταματήσουμε εκεί. Γιατί έχουμε αυτά τα εκατομμύρια ευρώ για τις ε, πρώτες επενδύσεις. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερο τι σκοπό έχετε για το μέλλον και θα ήθελα επίσης και να μου πείτε τι έγινε με τα αρχικά ποσά τα οποία επενδύθηκαν. Αν θέλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να γίνει στη συνέχεια μια στιγμή συζήτηση για το θέμα. Βεβαίω. Νομίζω ότι μπορούμε, όπως είπατε και εσείς, να δούμε την συνέχιση του Connecting Europe Facility, του μέσου συνδέοντα στην Ευρώπη, αλλά όπω είπε και ο συνάδελφο νωρίτερα, αξιοποιούμε και τη δυνατότητα τη τεχνολογία που προσφέρεται έξω από το Εύση ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Για τα 230 εκατομμύρια ευρώ βεβαίως έχουν αξιοποιηθεί ως μέσον προστασίας ένα χαρτοφυλάκιο έργων που παρατείνεται τώρα, επεκτείνεται έτσι ώστε να συμπεριλάβει και άλλα έργα υπό το ε, σύστημα εγγύσεων δανείων για τις μεταφορές έτσι εξασφαλίστε περισσότερη ε, ε, περισσότερος αντίκτυπος, μεγαλύτερη απήχηση δηλαδή των έργων αυτών που μπορούμε να ξεκινήσουμε με το ΕΦΣΙ και, από τα, και με τα ομόλογα έργου. Έχουμε καλύτερη δράση χαρτοφυλακίου και άρα περισσότερη αποτελεσματικότητα στο μέσον. Τα 237 εκατομμύρια ευρώ πάντως έχουν πλήρως αναπτυχθεί. Ο κύριος Τσέρνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και άλλα. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή για τα όσα μας εξήγησε, για την έκθεση αυτή που αναφορά τα ομόλογα έργο. Πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε για αυτόν τον οικονομικό έλεγχο από την Ernest Young. Βέβαια ε, κάπως ε, μαλάκωσε τις αξιολογίες κρίσης σε αυτή την ε, έκθεση. Γιατί έχουμε παρόλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θα ήθελα να μου δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία, κάποιες διευκρινήσεις για τα όσα συμπεράσματα έχετε εντάξει στην έκθεση και διαβάζοντας εγώ διαμορφώνω αρνητική άποψη για την εν λόγω πρωτοβουλία. Πρώτα-πρώτα, αυτό το οποίο ήδη γνωρίζαμε, ότι έχει την ίδια δομή όπως το πλάνο Γιούγκερ, όπως το Στατικό Ταμείο Επενδύσεων από πλευράς τεχνικής και από πλευράς ουσίας. Κατά κάποιο τρόπο, αν πραγματοποιήσουμε αν προχωρήσουν παράλληλα αυτές οι πρωτοβουλίες έχουμε αντιγραφή του, του, ενός από το άλλο. Άρα θα έχουμε άλλη μία από τα ίδια και τεχνικά και πολιτικά είναι εδώ να έχουμε διαφορετική ε, προσθεμένη αξία από ό,τι για το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Βέβαια έχουμε εδώ πέρα αυτές τις ε, διαρτικές επενδύσεις, έχουμε τη χρηματοδότηση που έχει με αυτόν τον τρόπο, την υποστήριξη δηλαδή της πρωτοβουλίας και η πρώτη μου σκέψη είναι ότι έχουμε εδώ χρηματοδότηση κάποιων έργων στις χώρες εκείνες οι οποίες δεν υπέστησαν αυτό το χτύπημα όσον αφορά ε, την κρίση σε επίπεδο επενδύσεων ε, υποδομής, αυτά τα οποία ξεκίνησαν το 2008, κάτι δηλαδή ε, αρνητικό το οποίο πρέπει να αναλυθεί. Επίσης, θα πρέπει να αναλύσουμε τα αριθμητικά στοιχεία για αυτά τα οποία εδώ έχετε υπολογίσει. Ας πούμε τους πολλαπλασιαστές που είναι τόσο υψηλοί στην έκθεση Ernest Young που λέει ότι ο, ποιος είναι ο στόχος και λέει ότι ο πόλεμο 15 με 20 είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει συνυπολογιστεί αλλά θα έχουμε τα νέα έργα. Πάντως μελετώντα αυτά τα στοιχεία διαπιστώνω ότι τα χρηματοδοτηθέντα έργα μας οδηγούν σε κάποιο είδους ε, ομόλογα έργων που φτάνουν τα 5 δις και μετά πάμε. Πόσα, πόσα εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 2-3 έργα τα οποία βρίσκονται εξελίξει, εξελίξη. Οπότε βλέπουμε ε, έχουμε αυτά τα 516 εκατομμύρια για το ομόλογα από την ΤΕΚΙ και άλλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα που είναι εγγυήσεις της ΕΤΕ οπότε Πάμε στα 5 δις που αφορούν την έκδοση των ομολόγων και επίσης 1,5 δις ε, από τον δημόσιο κορβανά και έχουμε τώρα 3,5 ως ε, συντελεστή προπλασιαστικού αποτελέσματος τώρα είναι κατακλείδη. Δεν πρόκειται έτσι να λυθεί το πρόβλημα των επενδύσεων στα έργα υποδομής, γιατί ένας ιδιώτης δεν πρόκειται να επενδύσει σε τέτοια έργα. Γιατί υπάρχει το ρίσκο της ε, κατασκευής. Αυτή είναι η φάση που εμπεριέχει το πιο μεγάλο κίνδυνο όταν δηλαδή δεν υπάρχουν ταμιακές ροές. Τότε ρισκάρει τα χρήματά του επενδυτής. Τέτοια εργαλεία επομένως πάρα πολύ συχνά δεν ωφελούν για να καλυφθεί ο σχετικός κίνδυνος. Αυτού του είδους τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται διακόπτει ο πρόεδρος. Κύριε Τζάνι, δεν πρόκειται περί ακρόασης. Μα είναι καλό να, είναι μελετημένοι και διαβασμένοι οι βουλευτές, αλλά τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Πρόκειται για τρία έργα, λέει ο κύριο Τζάνι, τα οποία είναι έργα Greenfield. Και έχουμε άλλα δύο τα οποία πέρασαν από χρηματοδότηση και άλλα τρία ε, αφορούν ε, ε, αυτά τα ομόλογα αλλά μιλάμε για λιγότερα από τα μισά που ήταν έργα τα οποία ενήχαν κάποιο κίνδυνο κατασκευής. Οπότε από αυτής της πλευράς πώς είναι να τον προχωρήσει αυτή η υπόθεση και να αποτελεί εγγύηση για τις επενδύσεις που θα γίνουν στην κατασκευή. Ήδη καλύψατε το είναι χρόνο χρόνο που θέλαμε να αναλώσουμε για απαντήσεις. Το επόμενο παρακαλώ είναι λίγο πιο σύντομος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής για την διεξοδική αυτή περιγραφή της εικόνας. Πολύ σύντομα θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες σκέψεις. Σε ποιο πεδίο κινούμαστε, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι εδώ δεν προχωρούμε σε μία αντιμετώπιση και από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών ή στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών, η οποία τελικά μας κάνει να χάνουμε τη γενικότερη εικόνα. Έχουμε αυτά τα ομόλογα έργου. Αποφασίσαμε και το ΕΦΣΕ, το σχέδιο Juncker. Τα έφτιαξε και ο κύριος Τσάνι νωρίτερα. Είναι αυτά τα πράγματα ε, λύσεις οι οποίες ε, προχωρούν παράλληλα, είναι αλληλένδετες έχει αποφασίσει η ΕΚΤ μια, μια πολιτική μηδενικών επιτοκίων. Με κάθε δυνατό μέτρο δηλαδή προσπαθεί να ενισχύσει την οικονομία. Ωστόσο ξέρουμε ότι έχει αναλάβει ε, χρέη μέχρι τα όρια του δυνατού ή του νοητού μέχρι τώρα. Επομένως, αυτό που μας λέτε είναι ότι πρέπει τα κράτη να αναλαμβάνουν ακόμη περισσότερα χρέη. Εδώ ακριβώ είναι το, άριο, το όριο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να καταστήσουμε ακόμη πιο περίπλοκα τα συστήματα μετακύληση του ε, χρέους ή τη χρηματοδότησης. Γιατί δεν έχουμε δει τίποτε άλλο από το 2007 και μετά, παρά μόνο μια μετακίνηση των ε, σχεδίων κατά τρόπον ώστε να ε, φτάνουν ακόμα και οι ειδικοί να λένε είναι τόσο αδιαφανή αυτά τα έργα, αυτά τα ομόλογα, αυτές οι λύσεις, που τελικά δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά πρέπει να τα υπογράφω. Αυτό δεν θα ήταν λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δυνανό. Πρόεδρε, ευχαριστώ όντως. Μάλλον είναι το ξαδελφάκι του σχεδίου Juncker το ομολόγο έργο, εκτός και αν το σχέδιο Juncker είναι το παιδί του ομολόγου έργου. Ενδιαφέρον πάντως να ενημερωθούμε αν αυτός ο ε, παράγοντας, παράγοντας μόχλευσης που ήταν η δόξα του σχεδίου Juncker είναι όντως αυτό που μας έχουν πει. Πάντως είναι πολύ κοντά και τα δύο στον ίδιο τομέα ή στους ίδιους τομείς κινούνται. Γνωστοί μεταφορές, ε, τηλεπικοινωνίες, ε, ίσως και περιβάλλον πιστεύω. Εκεί θα είναι χρήσιμο ασφαλώς να το κοιτάξουμε. Αλλά το ομόλογο έργου έχει βρει το business model του, πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, είναι λογικό να υπάρχουν δύο εργαλεία ταυτόσιμα ουσιαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος. Ωραία, κλείνω τον κατάλογο των αγοριτών για να δώσω την, την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να απαντήσει τουλάχιστον σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ναι, ευχαριστώ. Ξεκινώ με κάποιες διευκρινήσεις. Όταν ε, γίνεται λόγος για την ε, σχέση μεταξύ ομολόγων έργου και σχεδίου Juncker που έφυγε νωρίτερα δεν είναι συγκρίσιμα. Καταρχάς το ομόλογο έργο ήταν ένα πιλωτικό ε, έργο, ένα εγχείρημα το οποίο εισήχθη πριν από μερικά χρόνια για να δοκιμαστεί η αγορά των ομολόγων και το σχέδιο Juncker ξεκίνησε φέτος. Ο προπολογισμό στην αρχική πιλωτική φάση έχει ήδη δεσμευθεί και δαπανηθεί για το ομόλογο έργο. και όπως είδαμε, όπως είπαμε, ήδη υπάρχει υποστήριξη για τα φυστάμενα ομόλογα έργου και δεν θα χρειαστεί νέος προπολογισμό. Το ομόλογο έργο είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να προσφέρει το ΕΦΣΥ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε για το μέλλον. Είναι γιατί πρέπει να συνεχίσει το ΕΦΣΥ χωρίς να συνεχίσει το ομόλογο έργο. Τώρα έχουμε το εργαλείο Connecting Europe και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο διάβλους, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε το Connecting Europe κατά πάσα πιθανότητα και με ομόλογα έργου, χωρίς να έχω συγκεκριμένα παραδείγματα να σας δώσω για τα επόμενα έτη, αλλά ένα περιορισμένο προπολογισμό που έχουμε στο Connecting Europe θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε για να εστιαστούμε σε πιλωτικά, πειραματικά πρωτοπόρα ακόμη και ε, ε, υψηλής διακινδύνευσης προγράμματα για να ε, φτάσουμε να αξιοποιήσουμε δυνατότητες σε πιο, επίσημου, σε πιο επικίνδυνος ή υποδιακινδύνευση τομείς. Ενώ το ΕΦΣΙ θα έλεγα είναι ο παππούς του Project Bond. Έχει μια άλλη προσέγγιση δηλαδή και τελείως διαφορετικά κονδύλια. Και το Connecting Europe εστιάζεται μόνο σε έργα ερέσιμα επιλέξιμα. Ενώ το ΕΦΣΙ έχει πολύ ευρύτερη αντίληψη, καλύπτει κάθε τομέα επενδύσεων όπως άλλωστε αποφάσισε ο νομοθέτης. Θα ήθελα να πω σε σχέση με τα οικονομικά αυτά εργαλεία ότι η λογική δεν είναι ε, να προσπαθήσουμε να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά με χρέος τα κράτη-μέλη, αλλά να βρούμε λύσεις επενδύσεων για τις υποδομές. Αυτή είναι η προσπάθεια όλων μας βλέπουμε ότι είναι απαραίτητα αυτά τα ομόλογα, αυτά τα έργα μάλλον για όλες τις κοινότητες στην Ευρώπη και πρέπει ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο χρηματοδότησής τους με συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων πόρων κατά πάσα πιθανότητα, αλλά τώρα με αυτά τα μέσα προσπαθούμε να μεγενθύνουμε, να πολλαπλασιάσουμε όσο το δυνατόν τη διαθέσιμα ε, κονδύλια ε, τα ιδιωτική προελεύσεω περιορίζοντα το δυνατόν τη δέσμευση του δημοσίου. Και τώρα θα επιδώσω το λόγο και στον Νίκη να σα εξηγήσει λίγο περισσότερο τον παράγοντα τη μόχλευση. Ευχαριστώ. Όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα. Όταν μιλούμε για παράγοντα πολλαπλασιαστικό, μιλούμε για έναν λόγο μεταξύ του ποσού από ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που διαθέτουμε στην περίπτωση της πρωτοβουλίας πάλι, τα 230 δηλαδή αυτά εκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και, λόγω αυτού του ποσού, και τη συνολικής αξίας κόστους επενδύσεως για ένα έργο που καλύπτει, που υποστηρίζει το μέσον του ομολόγου έργου. Αυτή η μόχλευση λοιπόν τι λέει, ότι τα 237 εκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι διαθέσιμα ως δυνατότητα απώλεια σε ένα χαρτοφυλάκιο, εκεί που μπορεί δηλαδή να υποστηρίξει ένα, μπορεί να έχει ένα δευτερεύον χρέος ε, η ΕΤΕ, το οποίο ταυτόχρονα μπορεί να προσελκύσει άλλους επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως στην περίπτωση του ομολόγου έργου από την κεφαλαιοακή αγορά. Άρα το 3,4 δις επενδύσεων στο μεγαλύτερό τους μέρος, στο τεράστιο μερίδιο τους, είναι κονδύλια που επενδύει ο ιδιωτικός τομέας και δίκεφαλαιακή αγορά. Ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες. Ιδιωτικές. Άρα τι γίνεται σε σχέση με τα ποσά των ευρωπαϊκών πόρων αυτό που μπορεί να κάνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι μεγενθύνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Και χαίρομαι που μπορώ να συζητήσω το θέμα αυτό. Ε, ε, πολύ ευχαριστώ να συζητήσω το θέμα αυτό και δημερώσω ε, εάν χρειάζεται γιατί είναι αρκετά περίπλοκο αλλά πάντως αυτή είναι η βασική ιδέα και η πρωτοβουλία ομολόγων έργου και εύσου, εύση ακούστηκαν κάποια σχόλια και ο Τζόρτζο νομίζω τα άκουσε ότι μπορεί να είναι ο νόθος γιος του Εύση το ε, ομόλογο έργο. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ο υπερήφανος πατήρ. Γιατί, διότι η τεχνολογία την οποία μας εξασφάλισε σε όρους χρηματοοικονομικούς και χρήση ευρωπαϊκών πόρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα επιτρέψουν στην ΕΤΕ να αναλάβει ψηλότερο κίνδυνο και την προοπτική της ε, συγκέντρωσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα οφείλεται στο ομόλογο έργου και το Ευρωπαϊκό βέβαια Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ταυτόχρονα. <clears throat> Αυτό που εξήγησε και ο Τζόρτζ είναι ότι ήταν πιλωτική η δράση του ομολόγου έργου. Ήταν πρωτοπόρο και έτσι μπορέσαμε και για λόγους ε, σαφείς, ξεκάθαρους και αγαθούς που εξηγήσαμε στην αρχή, ένα έργο συγκεκριμένο με ενισχυόμενη την ε, υποστήριξη του πιστωτή και συγκεκριμένα την προσέλκυση, τη δυνατότητα προσέλκυσης και επανεξόδου σε αγορές ταξιδιωτικών ταμείων, ασφαλιστικών εταιριών κτλ. Στο ΕΦΣΥ έχουμε μεγαλύτερο, κλάδο, μεγαλύτερο φάσμα κλάδων, οικονομικών και μέσων. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι η αιτία αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο και έχουμε εργαλεία και στο χώρο της έκδοσης ε, χρεογράφων και στον χώρο του ε, χρέους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα και αυτό ακριβώς όπως υπόθηκε σημαίνει ότι μπορούμε με το Connecting Europe να συμπληρώσουμε αυτό που χρηματοδοτεί το ΕΦΣΥ. Πιστεύω να καλύπτονται τα ερωτήματα εκτός από αυτό ότι ο χρέους των κρατών μελών, της ανάληψης χρέους. Φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε και να συμφωνείτε ότι η ΕΤΕ διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα από, χάρη στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και προσφέρει υποστήριξη σε όλους τους μηχανισμούς, αλλά με ε, πλεονέκτημα σαφές, εφόσον και αυτό πράττει, εφαρμόσει τα δικά της ακριβή και αυστηρά κριτήρια. Μόνο δηλαδή οικονομικά υγιή ε, και τεχνικά βεβαίως, άρτια και περιβαλλοντικά αγαθά έργα μπορούν να ε, χρηματοδοτηθούν, να υποστηριχθούν από την ΕΤΕ. Μεταφέρεται δηλαδή ο κίνδυνος ε, από τον, δημόσιο, από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα και αυτό ακριβώς είναι ότι μπορούμε να καταφέρουμε και να εξασφαλίσουμε πολύ μεγαλύτερη απόδοση του χρήματος που θα δαπανίσουν οι δημόσιες αρχές. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και τους δύο από την ΕΤΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ καλή προσθέμενη αξία πάντως των παρουσιάσεων και βέβαια χάρη και στους συναδέλφους που τύπωσαν τις ερωτήσεις τους, υπενθυμίζονται μεταξύ ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ, έχει υπολογισμούς μόχλευσης πολύ ψηλότερους από αυτό που αναφέρεται εδώ. Εμείς έχουμε δει μέχρι 15-16 παράγοντα μόχλευσης. Με την ίδια βασική θεωρία από πίσω. Τώρα δεν ξέρω αν μπήκα και εγώ στον κατάλογο των αγορητών, αλλά πάντως δεν θα ανησυχούσα τόσο στο στάδιο που βρισκόμαστε. Σήμερα ακούμε ότι το ΕΦΣΥ έχει μπορέσει να φτάσει σε μόχληση 76 δις από την αγορά. Και είναι μόνο 6 μήνες που λειτουργεί το Ταμείο. Αυτά είχα να προσθέσω και εγώ. Μπορούμε όμως να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Α, να επιστρέψουμε στο σημείο 9 λοιπόν. Είναι για τον έλεγχο του Μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Είναι μια γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλία. Έχουμε την κυρία Τρούπαλ, η οποία είναι η συγγήτρια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είμαστε ε, σύντομοι, γιατί πραγματικά ε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Νομίζω πως ε, ακολουθούμε μια πολύ σαφή γραμμή. Θέλουμε νέους οριζόντιους κανόνες για να είναι πιο δίκαια και πολύ πιο διάφανη η σύνδεση των ομάδων εμπορογνωμόνων. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα ε, των ε, ημερησίων αποζημιώσεων, όπως επίσης και για το γεγονός πως θα πρέπει να γίνει δημόσια διαβούλευση με τους ΜΚΟ για τους νέους οριζόντους κανόνες, γιατί τότε μόνο πραγματικά θα έχουμε απευθυνθεί στο ευρωπαϊκό κοινό για να αποδείξουμε ότι υπάρχει πραγματική δέσμευση σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης νέων κανόνων να συζητήσουμε και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εδώ έχουμε εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας πω πως τα όσα ακούσαμε την τελευταία φορά ε, ήταν πως τους νέους οριζόντου κανόνες τους εξετάζει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και δεν περιμένει την έκθεση του Κοινοβουλίου. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν αποτελεί βέλτιστη πρακτική. Γιατί καλό θα ήταν την έκθεση του Κοινοβουλίου να την είχαν συμπεριλάβει ως τμήμα των νέων οριζόντιων κανόνων. Εάν πρόκειται πολύ σύντομα να καταθέσουν τους νέους κανόνες αυτούς ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε τουλάχιστον να ζητήσω να μας απαντήσει ο εκπρόσωπος Κομισιόν είναι ε, πρόθυμοι να διαβουλευτούν με τις ΚΟ μικρών στα πλαίσια των νέων οζόντιων κανόνων. Αυτό είναι ζωτική σημασία και μετά αφού απαντήσει ίσως κάνω και κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Τρούπελ. Ναι, όντως επιβεβαιώνει πως η Επιτροπή αυτή τη στιγμή προετοιμάζει τους νέους αναθεωρημένους οριζόντους κανόνες για τις ομάδες πυρογνωμόνων και είναι αυτοί οι κανόνες θα εστιάζουν, όπως αναμένει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι, στην διαφάνεια και στην ισορροπία. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις υπερεπαρκής για τους νέους οριζόντους κανόνες, οι οποίες θα στοχεύσουν στην αυξημένη και βελτιωμένη ισορροπία και διαφάνεια. Η κυρία Τρούπελ αναφέρθηκε στις ΜΚΟ. Εμείς θεωρούμε πως οι θέσεις και τα αιτήματα των ΜΚΟ σε μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί από το σχέδιο οριζόντιων κανόνων που σύντομα θα εγκρίνουμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2014 ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής όταν ε, έκανε μία ιδιαίτερη πρωτοβουλίας ε, έρευνα για το θέμα αυτό κάλεσε τις ΜΚΑ από την Ευρώπη να υποβάλουν απόψεις, παρατηρήσεις και σχόλια για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Το 60 με 70% των στοιχείων που υποβλήθηκαν εστάλησαν από ΜΚΑ προς το διαμεσολαβητή και αποτέλεσαν τμήμα των συστάσεων ε, της, Ευρω... διαμεσολαβήτριας που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς σχεδόν όλα αυτά τα αιτήματα τα συμπεριλάβαμε και επειδή συνεργαζόμαστε και πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και με τον εισηγητή εκεί, πρέπει να σας πω πως εκεί πιστεύουν πως οι νέοι κανόνες ακολουθούν μια ικανοποιητική πορεία σε σχέση με τις προσδοκίες και τα αιτήματα. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση, γιατί σε τεχνικό επίπεδο είμαστε πολύ προχωρημένοι και είμαστε έτοιμοι να εγκρίνουμε τους νέους κανόνες πολύ σύντομα Άρα λοιπόν δεν έχουμε στόχο να συμπεριλάβουμε μία ακόμα διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για τη διαβούλευση, μια και θεωρούμε πως τα αιτήματα τα σχετικά έχουν ήδη καλυφθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρούπελ. Απογοητεύομαι. Γιατί θεωρώ πως θα ήταν εξαιρετική ιδέα να γίνει αυτή η δημόσια διαβούλευση με, τους, με τις και όχι να εγκρίνουμε τους κανόνες χωρίς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για μένα αυτό σημαίνει πως εάν εγκρίνει τους νέους οι κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν υποβάλουμε εμεί στο Κοινοβούλιο την έκθεσή μας θα πρέπει να δούμε τους κανόνες αυτούς και να δούμε και πώς θα εφαρμοστούν και μετά αργότερα μέσα στη χρονιά να διαπιστώσουμε αν η εφαρμογή μας ικανοποιεί ή όχι και μετά να δούμε τι θα πράξουμε. Γιατί όντως υπάρχει και διαδικασία που μας επιτρέπει, αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Άλλος. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε το 9. The next one would be... Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, που είναι η αίτηση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης από τη Σουηδία. Ο κύριος Νεγκρέσκου που είναι δεν βρίσκεται εδώ. Η κυρία Γκαρδιά Σάβαλ που επρόκειτο να μας θα παρουσιάσει μόλις βγήκε από την αίθουσα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο. Προσέξτε κύριε Φερνάντες. Περνώ στα γρήγορα στο επόμενο που είναι κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Ο κύριος Νόβακοφ είναι και εκεί η Επιτροπής. Ο κύριος Φερνάντης ως συντονιστή του ΕΛΚ μας είπε πως θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση. bon, euh, κύριος Φερνάντες. Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά τεχνική βοήθεια. Στα πλαίσια του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μιλούμε για 360.000 ευρώ. τον κανονισμό δεν υπάρχουν προβλήματα τεχνικά ή νομικά. Ε, αυτά από πλευράς του συναδέλφου ο οποίος ήταν ο εισηγητής. Το μέγιστο ποσό θα πρέπει να είναι 0,5% όσον αφορά την τεχνική βοήθεια. Άρα, μιλούμε για 360.000 ευρώ. Κανένα πρόβλημα με το θέμα αυτό. Thank you. Any... ο πρόεδρος. Έχετε ερωτήσει κύριε Τόρβαλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε διαμέσου του κύριου Φερνάντες, τον εισηγητή τον κύριο Νόβακο θα πρέπει να παραδεχθούμε ε, βέβαια ότι για μένα δεν είναι ότι πιο αγαπημένο ή πιο δόκιμο να το θεωρώ αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, γιατί υπάρχουν και άλλα εργαλεία και άλλα μέσα τα οποία ε, βοηθούν στο να πιάσουν τόπο τα κοινωτικά χρήματα. Πάντω ε, είπε ο εισηγητής ότι χρειάζεται να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην προσταμινή αξία, επίσης στο πόσο εύχριστο είναι από του επιλέξιμου ε, τους δικαιούχου τέλο πάντων αυτό το ταμείο. Υπάρχει τώρα ένα θέμα με τα χρήματα και κατόπιν να δώσουμε την σκητάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας τα πει γιατί ακόμα και αν έχουμε εδώ συλλογή δεδομένων και αν χρησιμοποιούμε ξέρω εγώ πόσες ε, εργάσιμες ώρες για να πετύχουμε το στόχο μα, μπά και υπάρχει ε, κάποιο αποτέλεσμα γιατί ε, είπαμε ότι έχουμε την παγκοσμιοποίηση έχουμε κακή διαχείριση, άντι και κακοτυχία που χτυπά τις εταιρείε. Όμως αυτά τα δεδομένα ή αυτές οι δομικές αλλαγές, πώς θα καταλάβουμε, τι να σας πω, η πρώτη αντίδραση ενστικτόδηση είναι καταργήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζονται αυτά τα στοιχεία κανείς. Αυτό θα ήταν η σκεπτόδες αντίδραση μου. Πάντως, εάν μπορεί να έρθει η Κομισιόν και να μου δώσει μια ε, πιστική εξήγηση για το πόσο βοηθούν όλα αυτά τα στοιχεία, πόσο βοηθούν στο να πάει μπροστά η Ευρώπη, θα τη ήμουν ευγνώμων. Πάντως διατηρώ πολύ σοβαρές επιφυλάξεις, λέει ο κύριος Τόρβελτς, πρόεδρος. Άλλες παρατηρήσεις? Όχι, από ό,τι φαίνεται. Μήπως θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί τον ρόλο της. Εάν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να δώσω το λόγο εδώ στην παρακαθήμενη η οποία και έχει αναλάβει ε, τον φάκελο για τα θέματα ταμείου ποσμιοποίησης και να σας ενημερώσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομη απάντηση στην ερώτηση. Και νομίζω ότι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη θα σας δώσει την πλήρη απάντηση. Πρόκειται για κάποια στοιχεία ενημερωτικά τα οποία έχουμε συγκεντρώσει όσον αφορά το Ταμείο για την Μακροζημιοποίηση. Τα έχουμε σε αυτή τη βάση δεδομένων και είχαμε μια σειρά εκθέσεων πριν, τελευταία, πριν από λίγους μήνες που βασίζονται σε όλα αυτά και όλα αυτά υποβάλλονται στους αξιολογητές αυτοί που κάνουν την αξιολόγηση που θα τη στήσουμε και στο επόμενο θέμα της διάταξης. Οι εκθέσεις υπάρχουν ε, στο website της υπηρεσίας μας. Είναι τεράστια η βάση δεδομένων. Είναι το website του Ταμείου Κοσμιοποίησης. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα ενσωματώσουμε στο ΕΦΣΙ την βάση δεδομένων του Ταμείου Κοσμοποίησης που είναι πολύ πιο μεγάλο, πιο μεγάλη. Οπότε στο μέλλον θεωρούμε ότι θα μπορεί κανεί ε, να αναζητήσει τις πληροφορίες πολύ καλύτερα από την βάση δεδομένων του ΕΦΣΙ, την τράπεζα δεδομένων του ΕΦΣΙ. Πάντως, αν θέλετε, σας απαντώ και σε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, δεν βλέπω όμως άλλος να θέλει να υποβάλει ερώτηση. Ο Πρόεδρος. Βλέπω ικανοποιημένο τον κύριο Τόρβαλτς. Και προχωρούμε επομένως σε διάταξη. Έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες για την εν λόγω έκθεση που λύγει αύριο στις 6 η ώρα. Και στην Επιτροπή Αποσχόληση θα γίνει η ψηφοφορία. Σήμερα, σήμερα εμέλετο να γίνει. Και έγκριση του τελικού κειμένου στις 4 Απριλίου. Και στις 12 Απριλίου θα ψηφίσει η Βλομέλεια την εκθέση τώρα. Πάμε λίγο ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, όλα μέλη και πάμε πίσω τώρα στο 13 που είναι το Ταμείο Αποκοινοποίησης σε σχέση με την αίτηση της Σουηδίας και Αγκαρδία Θάμπαλ ε, αντί του κύριου Νεγκρέσκου του εισηγητού και να βγω ένα λεπτό από τη ε, συνεδρίαση. Εγώ εδώ έχω αντικαταστήσει τον κύριο Νεγκρέσκου. Έπεσε και αυτός από τη γρήπη που μας έχει πλέξει όλους. Ο κύριος Νεγκρέσκου θέλει να σας ενημερώσει πως μπροστά μας έχουμε ένα νέο αίτημα για το ταμείο αυτό που έχει υποβάλει η Σουηδία στις 18 Σεπτεμβρίου του 2015 και στο αίτημα αυτό είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ για 500 εργαζόμενους στη Βόλβο φορτηγά και άλλες επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από τις απολύσεις αυτές σε μια περιοχή της Βορείου Σουηδίας που δεν θα ε, δεν πρόκειται να σας πω το όνομά της γιατί νομίζω πως μπορώ να το προφέρω. Οι απολύσεις είναι λόγω της μειωμένης ζήτησης από την Κίνα η Volvo χρειάστηκε να μειώσει το προσωπικό της κατά 10%. Προφανώς η απώλεια αυτών των ε, θέσεων είναι κακό νέο, αλλά είναι πάντα χειρότερο όταν αυτό συμβαίνει σε περιοχές όπου λόγω γεωγραφικών ή κλιματικών συνθήκων η κατάσταση είναι πιο αρνητική για την εγκατάσταση καινούργιων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και αυτό συμβαίνει με αυτές τις απολύσεις που είχαν μεγαλύτερη επίπτωση ακόμα από ό,τι συνήθως στην περιοχή τους. Και γι' αυτό έχουμε το αίτημα για το ταμείο που ο εισηγητής θεωρεί πως είναι ε, απαραίτητο να δοθεί μια και όλα τα κριτήρια ε, τα οποία ισχύουν ε, πληρούνται. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σαβαρμά. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση γιατί δεν συμπεριέλαβε στο αίτημά της αυτό η Σουηδία. για έλεγχο και αναφορά τα κονδύλια τα σχετικά. Δυστυχώς δεν έχω ε, γνώση του θέματος. Το μόνο που έχω είναι τις σημειώσεις του κυρίου Μεγρέσκου που τελευταία στιγμή δεν θέλησα να σας παγιδεύσω. Ο λόγος που το θίγω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να μας απαντήσει. Νομίζω ότι είναι πάντω πάντως αυτές τι αιτήσει, σε αυτά τα αιτήματα, να συμπεριλαμβάνεται και αυτή η, η αίτηση. Οπότε θα πούμε πως ε, ως υποσημείωση πως δεν έχει ζητήσει τα σχετικά κονδύλια για την υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση η Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού λοιπόν με τη Φιλανδία, είναι αγορά ε, η, η οικονομία της αγοράς η Κίνα. Εσείς το λέτε για αστεία, αλλά αφού δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο, οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν. Σήμερα ή αύριο. Αύριο στις 6 το απόγευμα. 4 Απριλίου, τελική έκθεση και μετά 12 Απριλίου στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Και... και επειδή τα άλλα έχουν τελειώσει, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη έκθεση του κυρίου Ντένανο για την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014. Κύριε Σίγητα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντω μιλούμε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε εδώ έναν προπολογισμό 150 εκατομμυρίων το πολύ το χρόνο που μπορεί να χρηματοδοτήσει κατά 60% το κόστος ενός έργου και έτσι να βοηθήσει εκείνους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, να τους βοηθήσει να ξαναβρούν μια θέση εργασίας ή ενδεχομένως να φτιάξουν μια δική τους επιχείρηση. Πρόκειται πάνω απ' όλα για ένα εργαλείο αλληλεγγύης προς τον εργαζόμενο. Είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο. Μεταξύ 2007 και 2014, για να δώσω ένα παράδειγμα, 20 κράτη-μέλη έχουν καταθέσει για 134 ε, δράσεις που θα ωφελούσαν 120.000 εργαζομένους πάνω από 560 εκατομμύρια ευρώ. Λίγα λόγια έχω βάλει στο κείμενό μου. Περιμένω τις τροπολογίες. Είμαι αναγκασμένος να περιορίσω εγώ την έκταση. Ελπίζω να το βελτιώσουμε τις τροπολογίες και θέλουμε να κάνουμε και απολογισμό της λειτουργίας, τη πτυχή, τη δημοσιονομική βεβαίως Επιτροπή των Προϋπολογισμών, τη διάρθρωση με άλλα ταμεία όπως το κοινωνικό, άλλα μέσα κοινωνικής πολιτικής, κοινοτικής πολιτικής για υψηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών δράσεων και απασχολησιμότητα και απασχόληση την αξιοποίησή του και τον αντίκτυπο, τον πραγματικό αντίκτυπο για τον εργαζόμενο. Και σημειώνω ότι προσπαθούμε να κάνουμε και μία πρόβλεψη, δηλαδή να ε, αλλάξουμε ε, ουσία, κείμενα και ποσά για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ανάγκες. Ε, οι διορίες καταρχάς, οι προθεσμίες αναμονής είναι πολύ υψηλές, δεν είναι οι απαντήσεις, οι εξειδικευμένες ικανές να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα και διάφορες διαρθρωτικές ελλείψεις. Προκειμένου να δώσω κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα, συνάντησα διάφορους εταίρους του Ταμείου για τον Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, οπότε οι βασικοί παράγοντες ε, ε, αυτών των δύο θεμάτων ήταν η General Motors στο Βέλγιο και η άλλη μια στην Γαλλία και ήρθαμε σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι για αυτούς που απολύθηκαν και είπαμε ότι θα πρέπει να καλυφθούν από το Ταμείο αυτοί οι εργαζόμενοι. Και επίση είδαμε ότι ο Ζεπτοπλίστων είναι ευμενής η γνώμη που έχει διαμορφωθεί στους κόλπους του Ταμείου Οπότε αυτό το οποίο απαιτείται είναι ευελιξία και είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται επίσης και συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών ε, θεσμικών οργάνων, ιδίω των διαφθορτικών ταμείων, ούτω ώστε σήμερα να μπορούν τα κράτη-μέλη να συντονιστούν καλύτερα. Και βεβαίως θα ήθελα να δοθεί η παράταση της εξαίρεση για τα νίτς για μετά το 2017 αφού πρόκειται για ένα από τα κεκτημένα τα πιο σημαντικά του Ταμείου και απευθύνω και μία έκκληση να σκεφτούμε καλύτερα τη δυνατότητα για πρόληψη, για προληπτική δράση όσον αφορά την ε, αναμετατροπή τομέων δραστηριότητας γιατί μου λένε οι νέοι άνθρωποι με του οποίου έχω συναντηθεί ότι κάθε τομέα δραστηριότητα καταραίει ο ένα μετά τον άλλον καταραίουν οι τομεί δραστηριότητα, άρα πρέπει να κοιτάξουμε να προλαβαίνουμε τι εξελίξει. Το Ταμείο νομίζω πρέπει να προβλέπει περισσότερο, να κοιτάει πιο μακριά, να χρηματοδοτεί τομεακά, όπω είπα, προληπτικά. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει και τι μελέτε συνεπειών της παγκοσμιοποίησης ανατομέα και να κάνει δράσεις που θα βοηθήσουν τους πολίτες μας να προλάβουν τις ε, μετεξελίξεις ε, ανατομέα, τις τομεακές μετεξελίξεις και βέβαια να, προλάβουν επίσης, να προλάβουμε επίσης τις συνέπειες των απολειών, γιατί βέβαια το Ταμείο δεν έχει ρόλο μόνο να επουλώνει πληγές, αλλά πρέπει να προλαβαίνει κιόλας. Βεβαίω και πρέπει να υπουλώνει πληγέ, αλλά πρέπει να προλαβαίνει άλλου. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κύριο πνεύμα τη έκθεση. Ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Ζητεί κανεί το λόγο. Κυρία Γέτεμακη. Ευχαριστώ, όπω είπε και ο μιλητής μας. Πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε το εργαλείο αυτό εργαλείο αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους. Βεβαίως και θα πρέπει, κοιτάζοντας τη λεπτομέρεια, να συμπληρώσω ότι δεν δίνει μεγάλη προσθεμένη αξία, όπως είπε και ο συνάδελφος Νίλ Τούμπολ και το προηγούμενο θέμα. Σε κάποιες περιπτώσεις η αναδίπλωση ήταν μόνο 4%, ε, άρα είναι πολύ χαμηλή. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι έχει συμβολική αξία το Ταμείο για ορισμένου, αλλά θέλουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προσπαθώ να είμαι επικοδομητική λοιπόν και θα κάνω τις εξής παρατηρήσει. Πρώτον, θέλω ιδιαίτερα να δοθεί προσοχή στην ε, σπάνιδα των πόρων, που, μάλλον την απόκληση πόρων που ζητεί το Ταμείο και αυτών που διαθέτουν τα κράτη. Φαίνεται πως ο μέσος, το μέσο ποσοστό εκτέλεση προϋπολογισμού κινείται κάπου στο 50% και χρειάζεται βελτίωση. Άρα χρειάζεται καλύτερη ως προγραμματισμός και καλύτερη διαχείριση των έργων από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Πιστεύω ότι το ποσοστό συγχρηματοδότηση του 60% δεν πρέπει να αυξηθεί. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη τα ίδια να επενδύουν με δικούς τους πόρους και πρέπει να έχουν ενδιαφέρον να επιτύχουν τα σχέδια αυτά και όχι απλώς να τραβούν χρήμα που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ρημνά να χορηγήσει. Τρίτον, το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάνει κάποιους δημοσιονομικούς ελέγχους μεταξύ του Ταμείου και Εθνικών Ισολογισμών. Νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την επικάλυψη μεταξύ του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και του, ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό λοιπόν να μην υπάρχει επικάλυψη, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να υπάρξουν αποτελέσματα. το 4% του ποσοστού ανάπτυξης που είπα στην αρχή είναι πολύ χαμηλό. Ο κύριος Σαρβάμα, έχουμε ένα φιλανδικό ρητό. Ποτέ δύο φορές, πάντα τρεις. Και γι' αυτό ξαναστάω το λόγο γιατί έχω ακούσει τις επικρίσεις αυτές σε προηγούμενες συνεδριάσεις και θέλω υπο, οπωσδήποτε να υποστηρίζω τις επικρίσεις των συναδέλφων της Άλντε. Και ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κύριε Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ σύντομος. Όταν ρώτησα εγώ την κυβέρνηση γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ταμείο αυτό παρόλο που είχαμε επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω κρίσης, μας είπαν πως εντάξει, εμείς έχουμε την πολιτική συνοχής και μπορούμε τα χρήματα από το Ταμείο αυτής της Αλληλεγγύης να τα αφήσουμε για άλλα κράτη-μέλη. Και εάν ε, τελικά ξαναεκλεγεί η ίδια κυβέρνηση, νομίζω και τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα ίδια τα λέει. Δεν ζητά κανείς άλλος το λόγο λοιπόν. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο θα κάνω μια παρατήρηση. Είναι μάλλον περίεργο που θα πρέπει να περιμένει κανείς τις απολύσεις για να ξεκινήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, λόγω παγκοσμιοποίησης. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τις απολύσεις, θα πρέπει να μπορούμε να παρέμβουμε πιο πριν. Νομίζω ότι τελικά επαφίεται στην συνείδηση των κρατών μελών ε, και γι' αυτό το λόγο το αντιμετωπίζω στην... Ε, ε, το αντιμετωπίζω λίγο κοινικά, δηλαδή πολύ ωραία. Εμείς προσπαθούμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα του καταναλωτή, ε, φεύγουν και για να εγκατασταθούν σε άλλες επίρους οι επιχειρήσεις και για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας έχουμε αυτό το ταμείο, λέμε ότι εντάξει δεν μπορούσαμε να το προλάβουμε, αλλά νομίζω ότι τελικά ε, συμβαίνει το ίδιο και με τη μετανάστευση, γιατί πολλές από αυτές τις καταστάσεις θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί. Ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει να ε, εργαζόμαστε ανάντι. Τι σημαίνει αυτό πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο γρήγορα για να προσαρμόσουμε και να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις θέσεις απασχόλησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έκθεση λοιπόν συζητήθηκε σήμερα. Α, βλέπω που η κυρία, πως κυρία Γκάρθια Σάμπαλη ζητάει το λόγο. Με συγχωρείτε που ζήτησα το λόγο τελευταία στιγμή. Δεν μου φαίνεται δίκαιο από τη συζήτηση αυτή να δίνεται η εντύπωση πως ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν εξυπηρετεί τίποτα. Βέβαια, ξεκινά όταν οι υπόλοιπε πολιτικές έχουν αποτύχει και αυτό που θα πρέπει να πετύχουμε είναι να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική σφρίγιλη γιατί μιλούσαμε για τον αθέμητο ε, ανταγωνισμό από την Κίνα που μας επηρεάζει πολύ σήμερα το βιομηχανικό κλάδο της Ευρώπης και για παράδειγμα τη Χαλιβουργία, με ένα δική μου περιοχή έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίζουμε μέσω της βιομηχανικής πολιτικής, μέσω διαφορετικών πολιτικών, μέσω του ΕΚΤ για παράδειγμα. Και όταν όλα αυτά δεν έχουν ε, καταφέρει κάτι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη μικρή δυνατότητα βοήθειας που δεν είναι για να καθισχάσουμε τη συνείδησή μας αλλά για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι για να εκπαιδευτούν ε, πιο πολύ και να μπορέσουν να βρουν μια άλλη δουλειά. Είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεις ε, άλλη δουλειά, εντάξει δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς όποιος βγαίνει στην ανεργία δεν έχει και πολλές εγγυήσεις πως θα μπορέσει να ξαναβρει δουλειά. Οπότε νομίζω ότι ε, καλό είναι να λέμε πως το ταμείο αυτό έχει το συγκεκριμένο σκοπό που εξυπηρετεί, μην ζητάμε κάτι παραπάνω, είναι για όταν οι υπόλοιπε πολιτικές έχουν αποτύχει. Ναι. Αν μπορούσε όμως πριν τις απολύσεις να παρέμβει, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα ταμεία που το κάνουν αυτό. Το συγκεκριμένο ταμείο έχει στηθεί για τη φάση μετά. Είναι δηλαδή ο χαζαπλάς που βάζουμε πάνω στην πληγή. Αλλιώς είναι άλλες οι αποφάσεις και οι πολιτικές που θα πρέπει να λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη για να προλαμβάνουμε. Ακούω ανακρίβεις βεβαίω. Εντάξει, ότι πρέπει να γίνει καλύτερο προγραμματισμό, παρακολούθηση, να το δεχθώ, αλλά η... το ποσοστό αναδηλωση δεν είναι 4%, είναι 50%. Είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία, τα έχω δει. Είναι στοιχεία τη επιτροπή. 50% λοιπόν επαναπασχόλησης. Στον ίδιο τομέα και σε άλλους βέβαια. Αλλά εκεί πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή της αναδίπλωσης, της αν, ε, ανάληψης νέων δραστηριοτήτων και σε επίπεδο ε, Εδαφικό επίσης πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε πράγματα γιατί μπορεί να έχει κανείς κινητικότητα επαγγελματική αλλά όχι γεωγραφική σε επαγγελματικό επίπεδο μπορεί κανείς να αλλάξει ε, θέση εργασίας, αλλά να μην αλλάζει περιοχή εργασίας για διάφορους λόγους, γιατί είναι κατεστημένος εδώ και καιρό σε μια περιοχή, δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει τόσο εύκολα. Ένα ανθρώπινο δράμα κρύβεται πίσω από αυτό. Για τη συμμετοχή δε των ε, κρατών μελών, γιατί συμμετέχουν ανάλογα με την νομοθεσία τους βέβαια που τα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη, το δε ταμείο έχει παρέβαση πέραν αυτού που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Και επί της ουσίας, Πρόεδρε, γιατί το συζήτησαν πολλές φορές, το γνωρίζετε κι εσείς. Έχει το ταμείο αυτό ακόμα κάποια αξία, είπε και η κυρία Ζαπαλό, ότι πάνω απ' όλα έχει σημασία το ότι υπάρχει, αλλά έχει αξία και αποτελεί μια χτίδα ελπίδας για ορισμένους εργαζομένους, δεν πρέπει να τη σβήσουμε. Εάν λοιπόν μπορούσαμε να προβλέπουμε περισσότερο κάποιε μεταλλαγέ στου οικονομικού κλάδου, πίν του χάλιβα στην Ευρώπη, αν μπορούσαμε να προλάβουμε να δούμε ότι θα συμβεί, ίσω να μην βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε, να μελετήσουμε καλά τι παγκόσμιε αλλαγέ ε, και μεταλλάξει στην παγκόσμια οικονομία. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάιερ. Ε, συνάδελφοι. Νομίζω ότι αν μια επιχείρηση περιέρχεται σε δυσκολίες για λόγους διαχειριστικού ε, του management δηλαδή, υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Για λόγους παγκοσμιοποίησης μάλλον φταίει το management το ίδιο. Ε, υπάρχουν μηχανισμοί και στη δική μου την ε, περιοχή, στην Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, υπάρχουν μέσα, αλλά και είναι τελευταία λύσει το Ταμείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών τη παγκοσμιοποίηση, για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Σα το πω διαφορετικά. Φανταστείτε ένα ποδήλατο που έχει μόνο μία ρόδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να λέμε «Α, δεν λειτουργεί το ποδήλατο, να αφαιρέσουμε άλλη μία ρόδα». Μπορεί να είναι χαμηλό το ποσοστό της επαναπασχόλησης, το 50% που λέτε, να μας φαίνεται χαμηλό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το σταματήσουμε το Ταμείο. Δεν Μπορούμε να κοιτάξουμε τα, τα λάθη που υπάρχουν, τι ελλείψει που υπάρχουν σε επίπεδο αγορά-εργασία, το ότι δεν υπάρχει μια σωστή ε, ε επανεκπαίδευση. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε όμω χωρίς ε, περαιτέρω να σκεφτούμε την κατάσταση και πάνω απ' όλα χωρίς να, προβλ... και να είμαστε προσεκτικοί γιατί όταν επικρίνουμε κάποια ε, μέσα που έχουμε στη θέση μα θα πρέπει να είμαστε θέση να κάνουμε πληρέστερη ανάλυση. Μα ποιος είπε ότι θέλει να καταργηθεί. Απλώς πρέπει να ξέρουμε πότε θα διαθέτουμε τα κονδύλια. Παρακαλώ, Μαργάλ. Σύντομα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Κατιαθάμπαλ, εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων. Δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένο κανένα να διαλέξει, αλλά όπω και ο κύριο Ντενανό, καλύτερα πριν. Οπότε έχουμε αυτό το εργαλείο και ο κανονισμός πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει οι ίδιες οι επιχειρήσεις να προσφεύγουν στο σχετικό εργαλείο εκ των προτέρων. Και κατόπιν έχουμε τις άλλες προσπάθειες και τις ε, προτάσεις διάρθρωσες Οπότε να μην έχουμε στρεβλώσεις και αρνητικές επιπτώσεις. όπως ας πούμε την ε, παρέβαση νωρίς. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα ε, υπερλαμβάνεται η απόφαση γιατί ελήφθησαν όλα όσα έπρεπε. Ελήφθησαν όλα τα μέτρα που να όταν έπρεπε. Οπότε θα πρέπει να δούμε το με ποια διαδικασία καταλογίστηκαν ή χορηγήθηκαν αυτά τα κονδύλια. Και να δούμε και τις άλλες πολιτικές όμως που δεν μας απασχολούν για το συγκεκριμένο θέμα, τις πολιτικές επενδύσεων κλπ. Ωραία, ε, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτό το θέμα και οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν πριν την 23η Μαρτίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών 25 και 26 Απριλίου και στην ε, Ολομέλεια την 1η Ιουνίου. Και προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις ηλεκτρονικές ε, κάρτες στην συσκευή την οποία ψηφίζουμε για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν λειτουργεί. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας επί 25 ψήφων κλπ. Α, όχι, δεν λειτουργεί το δικό σας. Δεν έχω την κάρτα μου. Μπορώ να ψηφίζω μια ανάταση της χείρος μου. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Πρώτη ψηφοφορία. Έχουμε την έκθεση Καρδία Θάμπουλ. Και αφορά. Αλληλευτική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυροτανίας. Η συμφωνία είναι τετραετής. Ποιοι είναι υπέρ. Μπορείτε να ψήσετε δυνατά στους χείρος. Πρώτα ψηφίζουμε τη συμφωνία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα για την γνωμοδότηση της κυρίας Καρδιαθάμπολη. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 25 υπέρ και 26 με την κυρία Γιατεμάκη. Δύο κατά και τρεις αποχές. Έκθεση Μουρεσάν. Αλήθικη συμφωνία επίσης μεταξύ Λιβερίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της συμφωνίας. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές και για την γνωμοδότηση μου ρεσάν. Αν μας ψηφορία ψηφίζουμε. Πέρας. 24 συν για τον Μάγκη 25. 26. Τρεις αποχές, δύο ψηφίκατα. Κύριος Φερναντές. Κύριε Πρόεδρε, κάτι για την μεταφορά του 4. Πρόκειται για τρεις αληθικές συμφωνίες που έχουμε εδώ. Η με τη Μαυρτανία και δύο άλλες. Εδώ Μιλούμε για ένα παθηματικό 67,6 εκατομμύρια που αφορούν πιστώσεις υποχρεώσεων και 77 για πιστώσεις πληρωμών. C'est par appel nominal. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρο. Ψηφίζουμε. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. πέντε συν 1, 26. Δύο κατά δύο εποχέ. Για το άλλο μήμα, κύριε Ντεπρέ. Υπάρχει αίτηση μεταφορά. Α, υπάρχει. Πήγε πρώτα το λόγο ο κύριο ε, Φερνάντε. 150 εκατομμύρια είναι η μεταφορά που θα πρέπει να προέλθει από το αποθεματικό των κατεπηγόντων, κατεπηγούσης ε, βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται να καλύψει την ε, σειρακή κρίση και επίσης για να καλύψουμε τους πρόσφυγες σε Λίβανο και η Ιορδανία και γενικά τους εκτοπισμένους μέσα στην Συρία και στο Ιράκ. Θεωρούμε ότι είναι ένα ειδικό μέσο αυτό το αποθεματικό και έχουμε υποσχεθεί ότι αυτή η μεταφορά ε, θα γίνει. Το έχουμε υποσχεθεί από τον Οκτώβριο. Τώρα ψηφίζουμε, λέει ο Πρόεδρος, με ενωστική ψηφορία. Ψηφίζουμε. par 26 plus une 27. 26 συν Δύο κατά και μία αποχή. Monsieur Depré, il n'y a pas de demande de transfert sur les autres sections και τη συμμεταφορά κύριε Ντεπρέ για τα άλλα τμήματα. Κυρία Χόλμαγκερ για την πολιτική των ακινήτων. Οπότε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, λέει ο Πρόεδρος. Ουσιαστικά την ώρα που προβλεπόταν. Και τώρα κάνουμε μια λίγο λεπτή διακοπή, γιατί οι συνεδρία θα συνεχιστεί και κλεισμένων.